Okay, friends, we are unfortunately very few here. Uh, that's too bad. Uh, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι πολλοί παρόντες. Ε, κρίμα, αλλά δεν μπορώ να αναγκάσω και κανέναν να είναι παρόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς τροποποίησης. Ναι. Περνάμε στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης, ε, ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε διαπραγμάτευση με το με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με τον Eurofound και τον Σέντεφοπ. Και ο τέταρτο τριμερής διάλογος ε, πραγματοποιήθηκε χθε το βράδυ. Υπήρχαν πολλά τεχνικά σημεία, τα οποία τελικά συμφωνήθηκαν, αλλά τα βασικά πολιτικά θέματα εκκρεμούν ακόμα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν υπό την Αυστριακή Προεδρία. Ο επόμενος τριμερή διάλογος έχει, πραγματο... έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου. Δημιουργία κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που έχουν να κάνουν ε, με ε, άτομα και νοικοκυριά. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος πραγματοποιήθηκε 31 21 Ιουνίου και κατέληξε σε συμφωνία ανάμεσα στους συνομοθέτες. λαμβάνει η υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς ω προ του πόρου των στατιστικών ε, Ινστιτούτων. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί προς το παρόν για τις 11 Ιουλίου. Ε, ε, Έχουμε διερμηνία σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση. τις ε, συνθήκες υπό τι οποίε εργάζονται οι διερμηνείς. Παρακαλώ λοιπόν σημειώστε ότι... Σε περίπτωση που σε περίπτωση που δεν ε, καλύπτεται η συνεδρίαση αυτή, θα έχουμε διερμηνία μόνο στις ε, πέντε γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στην οποία είναι εμπλεγμένοι οι διερμηνείς. Οι διερμηνείς θα σας διαβάσουν το εξή μήνυμα. Βρισκόμαστε στην 24η μέρα των κινητοποιήσεων και ακόμα δεν έχουμε δει καμία αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Αντίθετα, ο Γενικό Γραμματέα κληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του. Στη σημερινή συνεδρίαση, πολλοί συναδελφοί μα από άλλε καμπίνε, όπω ακούσατε, έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Σε ένδειξη αλληλεγγύη, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασία όπω αρχικά προβλεπόταν. Ωστόσο, η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ στην προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Και τα τελευταία από τις τα τελευταία πρακτικά από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις των συντονιστών είναι στη διάθεσή σας, έτσι μπορείτε να διαβάσετε τι αποφασίστηκε. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 24ης Μαΐου δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Προχωράμε τότε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας και για όλες τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την ενσωμάτωση ε, υπηκών τρίτων χωρών. Και θα δώσω το λόγο στην Ελιάνα Ιλιανόβα που εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, είναι πάντα χαρά να βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση, ε, ακόμα και όταν είναι τόσο νωρί ε, το πρωί. Πριν ε, λίγο καιρό σα είχα μιλήσει για την εγγύηση για του νέου. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά να σα παρουσιάσω μια νέα έκθεσή μα. Δεν είναι έκθεση με συστάσεις, είναι ένα έγγραφο ενημερωτικό χωρίς συστάσεις. Θα είναι όμως χρήσιμο στη συζήτηση πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς λίγα λόγια. Η πρόσφατη αύξηση των ανθρώπων που ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στο επίκεντρο την ε, μεταναστευτική πολιτική και στο διάστημα 2014 έως 2017 σχεδόν 3,7 εκατομμύρια ανθρώπων ε, ζήτησαν άσυλο για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις φορές περισσότεροι από ότι την προηγούμενη τετραετία. Άλλοι έρχονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για σπουδές, για να ενωθούν πάλι με την οικογένειά τους για έρευνες. και συνολικά το 4% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Μια σειρά μελετών ε, έχει δείξει ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών ε, επιφέρει μακροπρόθεσμα ωφέλη οικονομικά και κοινωνικά για τις χώρες, αλλά η ενσωμάτωση των μεταναστών είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση εδώ είναι περιορισμένος, παρέχει κίνητρα και στηρίζει τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτών. Τι είναι λοιπόν ενσωμάτωση. Οι ανάγκες διαφόρων ειδών μεταναστών είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Και γι' αυτό απαιτείται δράση σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της παιδείας, της στέγασης, της απασχόλησης. Η ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελεί πρόκληση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ δεν υπάρχει επίσημος ορισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2004 το Συμβούλιο εκπώνησε 11 βασικές κοινέ αρχές για την πολιτική ενσωμάτωση που βλέπετε εδώ στην οθόνη. Όπως είπα στην αρχή, δεν θα δείτε ούτε συμπεράσματα ούτε συστάσεις. Πρόκειται για καθαρά ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο συνοψίζει τις δράσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενσωμάτωση των μεταναστών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε μία σύνοψη της παρουσίασης. Είναι πάρα πολύ σημαντική όμως, διότι παρουσιάζει τις 7 προκλήσεις που έχουμε εντοπίσει κατά τη διάρκεια των αναλύσεων μας. Η πρώτη έχει να κάνει με την ανάγκη μείωση των καθυστερήσεων. Σύμφωνα με τις μελέτες, όσο πιο γρήγορα ξεκινάει η ενσωμάτωση, τόσο πιο πιθανό είναι να πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο διακριτική ευχέρεια σχετικά με το πώ θα εφαρμόσουν την πολιτική στη χώρα του, που μπορεί να αποτελέσει λόγο για του ε, μετανάστε να μετακινηθούν από τη χώρα στην οποία ε, κατέφθασαν πρώτα σε άλλη χώρα, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την ενσωμάτωση. Άλλοι παράγοντες ε, είναι η καθυστέρηση διεκπαιρέωση των αιτήσεων, ενώ η δεύτερη πρόκληση είναι τα ίσα δικαιώματα και οι πολιτικές ε, κατά των διακρίσεων. Τα περισσότερα κράτη-μέλη καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μη γίνεται διάκριση εις βάρος των μεταναστών, ωστόσο σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017, το μεγαλύτερο ε, τμήμα των Ευρωπαίων πολιτών, ε, πάνω από το 50%, 54% για την ακρίβεια, έχουν ε, αρνητικό αίσθημα απέναντι στη μετανάστευση από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε δική μας έρευνα, τέσσερα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι η στάση του κράτους μέλους υποδοχής, ε, αν είναι αρνητική, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ενσωμάτωση. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η χρηματοδότηση και η αξιολόγηση των αναγκών. Δεν είναι σαφή τα πράγματα αυτή τη στιγμή, διότι διάφορα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση των μεταναστών με την αύξηση της μετανάστευσης ε, που είδαμε και που ανέφερα στην αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει 5 δισεκατομμύρια για τη μετανάστευση, εκ των οποίων 150 εκατομμύρια διατέθηκαν για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Αυτό το ποσό είναι σχετικά υψηλό, αλλά και μόνο το ΑΜΙΦ που είναι σχετικά μικρό διαρθρωτικό ταμείο ε, μας δίνει στοιχεία για τη μετανάστευση, τα οποία βέβαια μπορούμε να ελέγξουμε. Το συνολικό ποσό που δαπανούν τα κράτη-μέλη λοιπόν για την ενσωμάτωση των μεταναστών δεν είναι γνωστό, ούτε είναι γνωστός ο αριθμός των μεταναστών ε, που επωφελούνται. Κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΆΜΙΦ, ε, τα κράτη-μέλη είπαν ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια για την ενσωμάτωση των ταπανών. Οι πολιτικές ενσωμάτωσης επίσης πρέπει να περιλαμβάνουν ε, μια σωστή αξιολόγηση των αναγκών και θα πρέπει οι πόροι να διατίθονται την κατάλληλη στιγμή. Χωρίς όμως σωστό υπολογισμό των πόρων που απαιτούνται σε εθνικό επίπεδο, και ανάλυση του πώς ε, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώσει τις ανάγκες, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι αποτελεσματικές αυτές οι πολιτικές. Η τέταρτη πρόκληση συνδέεται με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που υιοθετήθηκε το 2016 αναφέρει τα βήματα που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενθαρρύνει όμως και τα κράτη-μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε επιπλέον μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν θα παρακολουθούνται στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κάτι που περιορίζει και τη δυνατότητά της ε, να παράσχει επιπλέον στήριξη στα κράτη-μέλη. Η επόμενη πρόκληση είναι να στηρίξουμε όλους τους, μετανάστες σε όλους τους τομείς πολιτικής. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εθνικές πολιτικές, άλλα κράτη-μέλη αναπτύσσουν μέτρα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ενώ άλλα κράτη-μέλη τα κάνουν όλα αυτά στο πλαίσιο άλλων πολιτικών. Πολλά κράτη-μέλη όμως δεν αναλαμβάνουν δράση σε σχέση με συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι οι απάτριδες ή οι νέοι μετανάστες. Επιπλέον εξετάσαμε τις εκθέσεις των ελεκτικών συνεδρίων όπου διαπιστώσαμε ελλείψεις στις πολιτικές ε, ένταξεις των κρατών μελών και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να στηρίζονται όλοι οι μετανάστες σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η έκτη πρόκληση που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έχει να κάνει με την διαθεσιμότητα δεδομένων. Είναι ένα πρόβλημα που βλέπουμε συχνά και σε άλλες πολιτικές. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν συγκεκριμένα τα αποτελέσματα στον τομέα των ε, μεταναστών. Δηλαδή, αν η χρηματοδότηση τους βοηθάει να ενσωματωθούν καλύτερα. Στην έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι δεν χρησιμοποιούνται δείκτες για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι εκθέσεις αυτές που μελετήσαμε επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ενσωμάτωσης και υπάρχουν ε, αδυναμίες στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών. Η παρακολούθηση των πολιτικών ε, με αξιόπιστα δεδομένα θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να προσαρμόζουν τις ε, πολιτικές τους ανάλογα με τις ανάγκες. Η έλλειψη σωστής πολιτικής, ε, ε, ε, σωστής παρακολούθησης μπορεί τελικά να εμποδίσει να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Η τελευταία πρόκληση έχει να κάνει με την περιπλοκότητα του τρόπου χρηματοδότησης. Ανακαλύψαμε ότι η νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να έχουν μηχανισμούς συντονισμού για να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη και να ε, περιορίσουν τις επικαλύψεις. Ωστόσο, η έρευνά μα ε, δείχνει ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τέτοιου μηχανισμού. Μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν εκδώσει κατευθυντήρε γραμμέ για τον συντονισμό και υπάρχει ανάγκη για ισχυρό ρόλο των κρατών μελών στην ε, διακυβέρνηση και στις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, υπολογίσαμε ότι πάνω από 400 διαφορετικοί οργανισμοί ε, συμμετέχουν στη διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των μεταναστών για το διάστημα 2014-2020 και επιπλέον 50 άλλους φορείς για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Χρειάζεται λοιπόν σωστό συντονισμός, διότι χωρίς σωστό συντονισμό υπάρχει κίνδυνος η πολυπλοκότητα αυτή να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές πολιτικές. Αυτά εν συντομία περιέχει το έγγραφό μας. Περιμένω να ακούσω παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω πολλούς ευρωβουλευτέ εδώ, αλλά ερωτήσει υπάρχουν από ό,τι βλέπω. Οπότε, παρακαλώ, κυρία Μάκεντάιρ πρώτα και μετά ο κύριος Χόρ. Και μετά η κυρία Γιονγκέριους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι από εδώ δύσκολα μπορώ να δω τις διαφάνειες. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ και αν μας τα δίνατε, μας τα στέλνατε και όλα αυτά τα, αυτό το PowerPoint, πολύ θα βοηθούσε. Λοιπόν, εγώ τώρα μιλάω βέβαια ως Βρετανή πολίτης. Η χώρα μου αγωνίζεται με αυτήν την ένταξη των μεταναστών εδώ και χρόνια. Και πρόκειται για πολιτική ανάγκη Όλα τα πολιτικά κόμματα δηλαδή πρέπει από κοινού να αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Μετά από το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα, διαπίστωσα ότι ξαφνικά υπήρξε μια αύξηση των εγκλημάτων μίσους. Πρόκειται βέβαια για ανθρώπους που χωρίς να ξέρουν καλά πως έχει η κατάσταση, ξαφνικά θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να εγκληματούν σε βάρος των μεταναστών. Εγώ είμαι από τα West Midlands. Εκεί ξεκίνησα μία οργάνωση που την ονόμασα West Midlands Together, μαζί. Και αυτό το έκανα με τους εργατικούς συναδέρφους. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι με τίποτα δεν πρόκειται για πρωτοβουλία ενός πολιτικού κόμματος. Όμως λέγοντας αυτό το μαζί θέλουμε να πούμε ότι μαζί είμαστε κατά κάθε μορφής εγκλημάτων ε, μίσους. έγινε αρκετά καλή δουλειά. Είχαμε μια διάσκεψη για τους νέους, όπου συγκεντρώθηκαν μαζί νέοι από διάφορα πολιτιστικά υπόβαθρα και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ θετικό και στηρίχτηκε. Όμως τι διαπίστωσε. Διαπίστωσε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ε, παράδειγμα για τη συνδυτοποίηση της ένταξης μεταναστών. Δεν χρησιμοποίησαμε άλλη χρηματοδότηση πέρα από χρήματα που μαζέψαμε σε εθελοντική βάση. Γιατί πρώτα απ' όλα γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά τα κονδύλια τα οποία μας αναφέρατε σήμερα. Αυτά που μας είπατε είναι πολύ ανασυχωτικό. Δηλαδή το ότι υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα, αλλά δεν υπάρχει αρκετός συντονισμός, ούτε και υπάρχει διαφήμιση αυτό των κονδυλίων. Δηλαδή, εμεί πώ θα ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα κονδύλια. Εγώ είμαι ευρωβουλευτή. Ε, πολύ θα ήθελα να το ξέρω ότι υπάρχουν και ότι θα μπορούσε να τα ζητήσει ο κόσμο αυτά τα χρήματα. Οπότε, συμφωνώ μαζί σα για το ότι θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και ενημέρωση. Έχω και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αναφερθήκατε σε πρόσθετα μέτρα, επιπλέον μέτρα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Δεύτερον, κάτι που με ανησυχεί πολύ, είναι η ένταξη των γυναικών. Ε, πολύ συχνά υπάρχει ο φραγμός της γλώσσας και συχνά οι γυναίκες βρίσκονται σπίτι, απομονωμένες, μόνες τους, περιορισμένες, ε, εξαιτία και κοινωνικών προδιαγραφών και δεν μπορούν να ενταχθούν μερικές φορές χρησιμοποιούν τα παιδιά τους που ξέρουν την τοπική γλώσσα ή ακόμα και τα εγγόνια τους, γιατί καμιά φορά τα παιδιά τους την ξέρουν. Και είναι τραγικό αυτό. Γιατί εμεί θέλουμε οι γυναίκες να μπορούν να παίξουν εξίσου ρόλο στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, να έχουν το ρόλο τους στην κοινωνία, όπως και οι άντρες. Χρειάζεται λοιπόν μια παραπάνω προσπάθεια για την ένταξη των γυναικών. Και αναρωτιέμαι αν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει και πού μας οδηγούν. Ευχαριστούμε, κύριο Χόρτσο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια και να σχολιάσω και να απαντήσω στο σχόλιο σας. Πρόκειται για τη διαμαρτυρία των διερμηνέων. Είμαι πολύ ενοχλημένος, είμαι εξοργισμένος από τον τρόπο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιδρά σε αυτή τη διαμαρτυρία. Λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόπος της δημοκρατίας. Η δημοκρατία και ο διάλογος είναι στο κέντρο της των εργασιών του Κοινοβουλίου. Δεν βλέπω ούτε διάλογο ούτε δημοκρατία εδώ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αυτών απαιτούν διάλογο και ζητούν συζητήσεις. Τους παραγνωρίζουν εδώ και καιρό και για μένα είναι απολύτως δυσάρεστη αυτή η κατάσταση. Με ενοχλεί βαθύτατα. Η Επιτροπή μας πιστεύω θα πρέπει να προβεί σε μία δήλωση ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται από την, Ευρωπα... από την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι διερμηνείς έτσι. Αυτό ως πρώτο σχόλιο. Για τις ερωτήσεις. Έχουμε εδώ ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο πρέπει να χειριστούμε με πολύ ε, προσεκτικό τρόπο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την ενσωμάτωση. Θα ήταν ουτοπικό να συζητούμε κάτι τέτοιο. Ερωτώ λοιπόν. Η παιδεία, η εκπαίδευση πώς μπορεί να προσφέρει, με τι μέτρα μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η εκπαίδευση να συμβάλλει στην ε, ε, ενσωμάτωση των μεταναστών. Μερικές φορές δίνεται η εντύπωση, ακούγεται ότι δεν θέλουν ε, να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία οι μετανάστες, ότι μπορεί να μην, να μην θέλουν να ενσωματωθούν γιατί έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους και λέτε ότι ίσως και το ίμιση να είναι αυτό το ποσοστό. Ε, σας έχει απασχολήσει το ενδεχόμενο να προσφερόταν στις χώρες αυτές με υποδομές που μπορούν να αναπτυχθούν, με δρόμους, με παιδικούς σταθμούς και άλλα και άλλα, ε, αυτή η δυνατότητα να ενισχυθεί η εκπαίδευση εκεί στις χώρες αυτές. Αλλά και άλλη τομείς, όχι μόνο η εκπαίδευση. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Πρέπει νομίζω να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτούς να μείνουν στις χώρες τους σε συνθήκες ειρήνης, να μην κινδυνεύουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί βλέπω ότι η μεταναστευτική μας πολιτική δεν φέρνει αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε λογικά μέτρα, χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα αυτών και από 1η Ιουλίου ξέρουμε ότι πρόκειται η καγκελάριος Μέρκελ να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα για τη μετανάστευση, πολύ ωραία, μένα, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την πολιτική στις χώρες αυτές. Κυρία Γιουγκέριος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, ευχαριστώ και για την έκθεση. Μας λέτε ουσιαστικά το που έχουμε κρίση με τη μετανάστευση και στην έκθεσή σας προτιμείτε να μας πείτε τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει καλύτερα από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Τώρα η κυρία Μακιντάιρ ομολόγησε ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα κονδύλια, έτσι. Και θα έλεγα ούτε κι εγώ το ήξερα. Μια ερώτηση για τη γραμματεία ίσως. Αυτά τα κονδύλια έμει. Ποια κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με τα κονδύλια αυτά, εμείς, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ποτέ στην επιτροπή μας μιλήσαμε για τα, αυτά τα κονδύλια τα ΕΜΗ. Α, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εντάξει, ωραία. Να, ένα παράδειγμα. Έλλειψης συντονισμού από την πλευρά μας. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα μια ερώτηση. Γιατί πολλά από τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε αποτελούν πρόκληση για τις χώρες μέλη. Και καλό θα ήταν να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα προκαλέσουμε συζήτηση σε επίπεδο χωρών μελών για τα ευρήματα της έκθεσής σας. Αυτό θα βοηθούσε νομίζω. Είμαι από την Ολλανδία εγώ. Και νομίζω ότι πήραμε τη λάθος απόφαση. Από φόβο θυμό της κοινωνίας. όσον αφορά προγράμματα για τους μετανάστες. Δηλαδή δεν θέλουμε πια να κάνουμε πολιτικές και προγράμματα ειδικά για τους μετανάστες. Ας πούμε για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. όχι τουλάχιστον ειδικά για τους μετανάστες. Και ίσως γι' αυτό σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν δεδομένα, γιατί μη θέλοντας να θυμώσουμε τον κόσμο επειδή έχουμε ειδικά προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών, ε, δεν ε, περιλαμβάνονται βέβαια σε καμιά στατιστική, είναι ένας φαύλος κύκλος. Τέλο πάντων, η πρώτη μου ερώτηση είναι, εσείς έχετε σχέδια για να προκαλέσετε αυτή τη συζήτηση σε επίπεδο χωρών μελών Έχετε προτάσεις για να προκαλέσετε δράσεις από εδώ στο εθνικό επίπεδο. Και κάτι ακόμα για το συντονισμό των κονδυλίων. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή υπάρχουν πολλές ε, οργανώσεις που εμπλέκονται σε όλα αυτά. Από την άλλη μεριά όμως, έχω την αίσθηση ότι αν πραγματικά θέλετε να εντάξετε στην κοινωνία σας μετανάστες, τότε είναι καλύτερα να αρχίσετε σε τοπικό επίπεδο. Να το παράδειγμα που έδωσε η συνάδελφος ήταν πολύ ωραίο. Ή, εν πάση να προκαλέσετε την ε, συμμετοχή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να αναλάβει και αυτή το δικό της μερίδιο για προγράμματα κατάρτισης κλπ. Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος όταν λέτε ότι χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό τελικά η οργάνωση να γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε ή μήπως ανάποδο, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί πάρα πολλοί συμμετέχουν σε θελοντική βάση για να βοηθήσουν στις διάφορες κοινωνίες μας. Αν λέτε 400-500 νεκροί είναι πάρα πολύ, Και τελικά μήπω αυτού του είδους η οργάνωση δεν βοηθάει. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Σε σχέση ακριβώς με αυτά που μόλις είπε η κυρία Γιονγκιάριος, ακριβώς αυτή η ένταξη από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω, και εμένα με απασχολεί. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή αυτή Απασχόλησης, η Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Απασχόλησης έχει αρμοδιότητα, όπως και κοινοβουλευτικέ επιτροπές, να δείξουν συγκεκριμένους τρόπους προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα σε κάποιες χώρες μέλη και που έχουν να κάνουν με την ένταξη ή την μη ένταξη τελικά των μεταναστών. Και βέβαια θα σας μιλήσω για τη δικιά μου περίπτωση, τη δικιά μου χώρα. Στη Σουηδία είμαστε 10 εκατομμύρια. Και πήραμε σχεδόν ένα εκατομμύριο μετανάστες, σε πρόσφυγες μάλλον, σε ένα ε, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάποιοι φύγαν και πήγαν αλλού, αλλά πάρα πολλοί έχουν παραμείνει στη Σουηδία. Και θα ζήσουν στη Σουηδία. Τουλάχιστον αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει οι αρχές σε πολιτικό επίπεδο. Συμφωνούν σε αυτό. Άρα πρέπει να βρούμε λύσεις που δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μια κρίση που διαρκεί πέντε μήνες ή πέντε χρόνια. Πρόκειται πραγματικά για την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Με πολιτική συνένεση λοιπόν στη Σουηδία, ευρεία πολιτική συνένεση, ένα μεγάλο μέρος της ένταξης αυτής έχει να κάνει με το πώς οι άνθρωποι αυτοί που προέρχονται από τελείως διαφορετικά υπόβαθρα συνήθως θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Άρα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να καταστεί δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί μη γνωρίζοντας ούτε λέξεις σου ειδικά, να μπορούν παρόλα αυτά να βρεθούν σε κάποιο χώρο εργασίας, να συνεργαστούν με άλλους εργαζόμενους και να έχουν και την δυνατότητα να μάθουν και τη γλώσσα, να τη διδαχτούν. Στη Σουδία λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργαδότες και εργαζόμενοι, κατέληξαν σε συμφωνία ότι θα διαχειριστούν το ζήτημα αυτό από κοινού. Το πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση εννοείται συμμετέχει, αλλά είναι οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι τελικά αποφάσισαν πώς θα ενταχθούν οι πρόσφυγες μακροπρόθεσμα μέσα από την εργασία τους στην Σουηδική Αγορά Εργασίας. Βέβαια και είναι περίπλοκο και μερικές φορές σε κάποιους κλάδους, σε κάποιες περιοχές της χώρας, αλλού πάει καλά το πράγμα, αλλού υπάρχουν προβλήματα. Πάντως θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και ελπίζω στη Σουηδία τουλάχιστον να έχουμε θετικά αποτελέσματα γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλες χώρες μέλη. Εμείς εδώ μιλάμε τόσο πολύ για το πώς θα εντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς, ματώνει η καρδιά μας. Δεν είμαστε ρατσιστές, εντάξει υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ χωρών μελών, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις. Να μιλάμε περισσότερο και να καταλήγουμε σε έργα. Οι κοινωνικοί εταίροι λοιπόν στη Σουηδία, ίσω και σε άλλε χώρε μέλη, κατέληξαν σε λύση. Αν έχει δουλειά, είναι καλό. Βλέπουν τα παιδιά σου, ότι οι γονεί του έχουν κάποια καθήκοντα έξω από το σπίτι, δουλεύουν. Είναι καλό γιατί έτσι μαθαίνει πιο εύκολα τη γλώσσα. Στην πράξη, μέσω τη δουλειά σου. Και βέβαια κερδίζει και χρήματα. Και αυτό σου προσφέρει αξιοπρέπεια και σου δίνει και δύναμη. Νιώθεις πιο δυνατός. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση σίγουρα. Πάντως η ένταξη των προσφύγων δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σε λίγα χρόνια, σε τρία χρόνια το έχουμε λύσει. Όχι, θα πάρει πολλά χρόνια. Τώρα, έρχομαι στην ερώτησή μου. Έχετε προτάσεις στην πράξη για το τι να κάνουμε, έναν κατάλογο to do. Ε, σίγουρα υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, διαφορετικές καταστάσεις. Όμως Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει ένας τέτοιος κατάλογος στον οποίο να μπορούν να συμβουλευτούν όλοι, κάθε κοινότητα, κάθε χώρα, ώστε να τον μελετήσει τον κατάλογο, να τον εξετάσει και να αποφασίσει τι από αυτά μπορεί να κάνει και τι από αυτά δεν μπορεί να κάνει. Υπάρχουν χώρες μέλη που τα κατάφεραν, είτε σε μικρή κλίμακα είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και πρέπει να ξέρουμε τι κάναν και πέτυχαν, τι αλλαγές έκαναν και πώς κατάφεραν να έχουν αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, αλλά το μυαλό μας να το κατευθύνουμε σε πρακτικές λύσεις. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα χρήσιμα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις αυτές. Ας αρχίσω από το τέλος. Όντως, η ένταξη είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα και όχι εύκολο. Παίρνει χρόνο να πετύχουμε την ένταξη και μετά να μετρήσουμε και τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα λόγο που δεν κάναμε ειδική έκθεση, παρόλο που πρέπει να ομολογήσω, στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή μα. θέλαμε να έχουμε μια έκθεση, αλλά μετά διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τόσο περιορισμένα, δεν είναι αρκετά διαθέσιμα, οπότε ήταν καλύτερα να ξεκινήσουμε ε, καλύτερα με μια τέτοια παρουσίαση μικρής κλίμακας και να δούμε σιγά σιγά τι παραπάνω στοιχεία έχουμε. Λοιπόν, αρχίζω από το τέλος, έτσι ρωτάτε. Ε, τι κατάλογο θα μπορούσαμε να συντάξουμε με πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αρχίζουμε με το πρώτο βήμα, που είναι να κατανοήσουμε την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, να εντοπίσουμε τις προκλήσεις και έτσι να προκαλέσουμε συζήτηση, όπως είπε και η κυρία Γιονγκέριους. Πώς θα προκαλέσουμε τη συζήτηση στις χώρες μέλη. Αυτό είναι κάτι που αποτελεί μέρος των όσων κάνουμε. Δηλαδή πάμε στις χώρες μέλη, ε, μπαίνουμε σε συζητήσεις και όποιος μας καλέσει, βεβαίως και πάμε, αν μας καλέσετε ευχαρίστω. Πρόκειται για μια πολιτική που δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, το είπατε κι εσείς. Ό,τι γίνεται, γίνεται σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Και τα μέτρα αποκρίνονται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Θα έρθω όμως τώρα στην ε, πρώτη ερώτηση και τα σχόλια της κυρίας Μακεντάιρ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα προφανές παράδειγμα και επιχείρημα που ενισχύει ακριβώς τα δικά μας ευρήματα, πώς θα αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχει αυτό το μίσος, το έγκλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι κάτι που κι εμείς έχουμε εντοπίσει. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, είναι προφανές και είναι μια σημαντική δυσκολία, διότι αν δεν γνωρίζετε πόσα χρήματα χρειάζεστε, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσετε και να έχετε αποτελέσματα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά πρέπει τα αποτελέσματα να μετρώνται. Αλλιώς το πιο πιθανό είναι να μην τα καταφέρετε. Οπότε ναι, χρειάζεται φυσικά ε, καλύτερο συντονισμός και καλύτερη ενημέρωση για τα διαθέσιμα κονδύλια. Επιπλέον ε, μέτρα με ρωτάτε. Κατάρτιση, εκπαίδευση, που όσο πιο γρήγορα αρχίσουν, τόσο το καλύτερο. Γλωσσικά μαθήματα, ε, μαθήματα επιχειρηματικότητας, ένταξη γυναικών. Βεβαίω αυτά δεν είναι βέβαια για όλε τι χώρε. Το είπατε κι εσεί κυρία Πρόεδρε, στη χώρα σας άρχισαν αλλιώ τα πράγματα. Πρώτα δουλειά και μετά γλωσσική κατάρτιση. Δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή. Στην κάθε χώρα πρέπει να δούμε τι θα λειτουργήσει καλύτερα. Η ανταλλαγή πάντως βέλτιστων πρακτικών, κάτι που κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα είναι κάτι που βοηθάει. Έτσι μαθαίνουμε ένας από τον άλλον. Τα δεδομένα, όπως σας είπα, είναι πολύ περιορισμένα για να μετρήσουμε, όπως με ρωτήσατε, ποια είναι τα αποτελέσματα των προσπαθειών που γίνονται για την ένταξη των γυναικών, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να σας πω για καμία ομάδα μάλιστα ε, βάλω των ατόμων. Ούτε καν τα συνολικά δεδομένα δεν υπάρχουν καλά-καλά. Οπότε πόσο μάλλον για την περίπτωση των γυναικών. Ελπίζουμε, μια που είμαστε σε μια διαδικασία που παίρνει χρόνο, ελπίζω αργότερα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Τι άλλα σχόλια τώρα κάνατε για την ένταξη. Ναι, είναι μια διαδικασία αμφίδρομη. Συμφωνώ με αυτό. Το λέμε και εμείς στην εκθεσή μας. Ότι υπάρχουν δύο πλευρές στην ένταξη. Ο ένα είναι που αποδέχεται την ένταξη και ο άλλο είναι που την προσφέρει. Άρα πρέπει να θέλεις να ενταχθείς για να ενταχθείς, έτσι. Συζητώντα γενικά τώρα την μετανάστευση, εμείς λέμε ότι είναι μέρος της ένταξης, το λέμε στην αρχή, ότι καταλήγουμε στην ένταξη μετά από μια συνολική διαδικασία και αρκετά περίπλοκη μάλιστα. Τώρα. Α, για το πώς θα γίνει αυτό, από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Πολύ καλό σχόλιο και κάπως με προκαλείτε εδώ, αλλά καλά κάνετε. Δεν έχω να σας δώσω συστάσεις ή συνταγές, γιατί όπως σας είπα δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι σαφώς ο εντοπισμός των προκλήσεων για καλύτερο συντονισμό δεν σημαίνει ότι ζητάμε περισσότερη εναρμόνιση ή κοινέ πολιτικές, όχι. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις Πρέπει να καταλάβουμε καλά ποια είναι τα είδη χρηματοδότησης για να αποφύγουμε ένα μέτρο, για παράδειγμα, να χρηματοδοτείται, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε καλά-καλά από τι κονδύλια, μπορεί να χρηματοδοτείται και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ κάποιο άλλο καθόλου να μην ε, υπάρχουν τέτοιε επικαλύψει για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε, εγώ δεν θα έλεγα από πάνω προ τα κάτω ή από κάτω προ τα πάνω. Δεν έχω να σα κάνω τέτοια σύσταση, αλλά καλύτερο συντονισμό να έχουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το γενικότερο πλαίσιο, τη μεγάλη εικόνα να έχουμε υπόψη μα για να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. Και θα τελειώσω με κάτι που είπατε εσεί, κυρία Πρόεδρε. Το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για έκθεση με συστάσει, όχι. Όμως πρέπει να σας πω έξω από αυτό το κείμενο ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι ο τελικός στόχος. Γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, ε, μαθαίνουν τη γλώσσα, ετάσσονται στην κοινωνία. Γιατί, για να ενταχθούν και στην αγορά εργασίας. Και τέλος κάτι από το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε, είναι βέβαια πολύ νωρίς για να σας το υποσχεθώ, αλλά αν έχουμε κάποια άλλη ακρόαση γι' αυτό, μια σύσταση θα ήταν αυτό που είπατε κι εσείς, λιγότερα λόγια, περισσότερη δράση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να συζητήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, στις 10 η ώρα θα ψηφίσουμε. Θα περιμένουμε λοιπόν 6 λεπτά. Μήπως έρθουν και άλλοι ευρωβουλευτές. 5-6 λεπτά κουβεντούλα λοιπόν. Okay, we shall vote, we are not... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε. Δεν είμαστε πολλοί παρόντες. Αλλά φαντάζομαι ότι οι λοιποί απόντες έχουν άλλες υποχρεώσεις. Ξεκινώ με την γνωμοδότηση. Πανευρωπαϊκό προϊόντα συνταξιοδότησης. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τίτλος πρώτος τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 170 κατά πίπτη και πάμε και στην 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 173 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 174 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 175 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 176 υπέρ κατά αποχές Καταπίπτει λοιπόν. Καλό σας ε, το ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. «22 ψήφοι υπέρ» και άρα είναι απλά τα πράγματα και Πάμε στην 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθή. 179 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 180 υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύουμε την 180. Δεν ήταν απολύτως σαφές το αποτέλεσμα. Αρχή φορεία, πέρασε. Και εγκρίνεται 21, 21 ψήφους υπέρ και 17 κατά. 181 τώρα υπέρ, κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε και την 181. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. 182 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 183, 184, 185, 186 καταπίπτουν όλες και πάμε στην 187 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 188 καταπίπτει, 189 καταπίπτει. 190, 191, 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες και πάμε στην 196 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Πάμε μέχρι τη 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 203 καταπίπτει. 204 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ας επαληθεύσουμε τη 204, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Με 22 ψήφους εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 206 καταπίπτει, 207 καταπίπτει, 208, 9. Στη 210 υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. 211 καταπίπτει. 212 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε 212. Πέρας στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους 213. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε τη 213. Πέρας. Απερίφθη με 21 ψήφους. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ε, μάλλον τροπολογία 219 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 200, ε, η συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. 224 καταπίπτει. 225 υπέρ. 225 υπέρ κατά Αποχές απεριφθεί. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές απεριφθεί. 228-229 καταπίπτουν. 230 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απερίφθη. 231 ένα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 232 μαζί με την 233 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 234 υπέρ κατά απόχες απερίφθη 235 υπέρ κατά αποχές Απερίφθη. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές και λέω ότι απερίφθη, αλλά ας επαληθεύσουμε τη 236. Απερίφθη. 18 ψήφι κατά. 237 μαζί με τη 238 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 241 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Διακόσια σαράντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. και εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. ...246 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε τη 248. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 21 ψήφους. Υπέρ. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 251. Πέρας 26 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 252 και όχι. «252 υπέρ» κατά αποχές απερίφθη. 253 καταπίπτει. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, ε, απερίφθη, συγγνώμη. 254 υπέρ κατά αποχές επερίφθη ή 255 κατά πιεπτή 260 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε τη 260. Πέρας. 22 ψήφι υπέρ. 261 καταπίπτει. 262 Υπέρ. Κατά. Αποχές περίφθει. Επαληθεύουμε λοιπόν τη 262. Αρχίζει η ψηφοφορία. Με 21 ψήφους υπέρ εγκρίνεται. 263 καταπίπτει. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 283 υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε τη 283. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρασε. Με δύο ψήφους διαφορά εγκρίνεται. 285 λέει πρόεδρος, όχι καταπίπτει. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 290 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται μάλλον. 12 καταπίπτει. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 297 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 297 επαληθεύουμε πέρας εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ η επόμενη καταπίπτει πάμε στην 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 301 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 302 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 303 καταπίπτει, 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, amendment 306. Ε, 306 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 306. And the vote is now closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 36 ψήφους. 307 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 308. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, the vote is now closed. πέρα εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Η 309 καταπίπτει. 310 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 311 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 312 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 316 και 317 ε, καταπίπτουν. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ή ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 372 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 373 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ. Κατά επαλήθευση της 375. Άρχεται η ψηφοφορία. And uh, it's now closed. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Υπέρ. 376. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 377. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β, Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 394, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. Επαλήθευση. Της 394 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. 396 υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση 396. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με πλειοψηφία δύο ψήφων. 397 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 401 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 404 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 404 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 ψήφους κατά. 405 υπέρ. Ε, κατά ε, αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 406. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται ε, με 19 ψήφους κατά, κατά δύο ψήφους δηλαδή. 407 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 409 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 410 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 413 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 413. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 417 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 418 καταπίπτει, 419 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 420 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 420. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. S&D έχουμε μία ψήφο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. εγκρίνεται με πλειοψηφία δύο ψήφων. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 422. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με πλειοψηφία μίας ψήφου. Τροπολογία 423 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 424 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 426 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 427 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 428 καταπίπτει. 429 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 430 και 431 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 432 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 433 καταπίπτει. 434, όχι δεν καταπίπτει. Και η, και 434 καταπίπτει. 435. Ψηφίζουμε 435 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 435. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά δύο ψήφους. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Λυπάμαι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 19. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. Τροπολογία 20. 437. Όχι. Μόνο την 20 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 437 καταπίπτει. Και η 438. Περνάμε στην 439 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 448 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι, καταπίπτει. Εφόσον ε, εγκρίθηκε η 448, όχι, απορρίφθηκε, άρα εντάξει. Τροπολογία 22 απορρίπτεται. Όχι, 22 εγκρίθηκε. Η 448 απορρίφθηκε. Η 22 εγκρίθηκε. Περνάμε στην 452 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 453. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 453. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. «455» είναι η επόμενη τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 460 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 461 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 479 υπέρ, κατά, επαλήθευση, 479, άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is now closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 478 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 478. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. 481 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται νομίζω. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πάλι. 482 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω καλύτερα να επαληθεύσουμε 482 άρχεται η ψηφοφορία Πέρα της ψηφοφορίες. εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. 483 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 484 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 484 λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη. 484 λέει πάλι η πρόεδρος but uh, Yes. Yes, we have already voted on 483. Ψηφίσαμε ήδη τις 483 και 484. Προχωράμε στην 485 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 485. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay, we stop there. And it is carried by 20 votes. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ. 486 καταπίπτει. 487 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 489 καταπίπτει. 490 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τετρακόσια ενενήντα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 491. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 492 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 492. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. 493 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 495. Καταπίπτει. Ωραία. 494 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 497. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 498. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 499. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 500. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 501. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 502 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 503. Είναι η ίδια με την επόμενη. Όχι. 503. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 504. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 505 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 506 μαζί ή όχι. Όχι, 506 μόνη της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 507 καταπίπτει 508 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 509 καταπίπτει. 510 τώρα υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 511 εκπίπτει. Τροπολογία 27 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30. Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 21 ψήφοι υπέρ. Τώρα. Συμβαστική α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 2. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε 25 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 35 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια σας. Α, έτσι. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 3 παρακαλώ. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 37 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 23 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 38 τώρα, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 38. Ναι. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε με δύο ψήφους φορά Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε για την τροπολογία 42 ηλεκτρονικά. <coughs> Πέρα στις ψηφοφορίες και απορρίφθηκε. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 47 παρακαλώ, ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 24 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 50 τώρα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52, 53 και 50... Όχι, μόνο 52 και 53 μαζί υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά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 Τέλος. Απορρίφθηκε. 21 ψήφι κατά. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Α, να ελέγξουμε. Ωραία, θα ελέγξουμε. Εντάξει. 63. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 65 με την 66 μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, α, κατά πίπτη μου λένε. Ωραία. Τροπολογία 70 τότε. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 70. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Με τέσσερις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 79. 79 Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81. Υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύσκολο να... Πολλά εγκρίνεται νομίζω. 84. Α, καταπίπτει. Αφού εγκρίθηκε η 83. Τροπολογία 85 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη. Όχι, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρο. Τροπολογία 90, Κατά πίπτη. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λέτε. Τροπολογία 7. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία. Ναι, εγκριθήκε με 39 ψήφους. Υπέρ, δεν απορρίπτεται προφανώς. Καλά, μήπως διάλειμμα όταν έχουμε ήδη ψηφίσει το σύνορα. το τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 πίπτη. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 101 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Η 102 καταπίπτει. Τροπολογία 103 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Για την 107 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. 107. Πέρας. Απορρίφθηκε. 108 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και αυτήν, έτσι κι αλλιώς πριν ήταν ισοψηφία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά 108. Πέρας. Και εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 109. Υπέρ. Κατά. να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έτσι κι το αποτέλεσμα είναι πάντα τόσο τσιμα-τσιμα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 109. Τέλος. Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 110. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, Α, να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική G, Z. Ψηφίστε παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία και εγκρίθηκε 22 ψήφι υπέρ. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 117 ηλεκτρονικά μπορείτε να ψηφίσετε. Εγκρίθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 όχι 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 126, δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη, πρώτο τμήμα, πρώτο, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, δεν το έχετε βρει. Είμαστε στην τροπολογία 126, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 πάντα δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα. πέρα της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. Τροπολογία 127. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 127 ελέγχουμε, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, παρακαλώ, ησυχία τώρα που ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Τα πηγαδάκια είναι για αργότερα. Τροπολογία 38 καταπίπτει, τροπολογία 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 και 145 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 146 κατά πίπτη, 147 τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την 147 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 154 υπέρ, 154 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την 156. Ωραία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος, απορριφθήκε. 20 ψήφοι κατά. Τροπολογία 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 158 πρώτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ. Ε, τώρα 158 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ. Κατά. Τρο... Αποχές απορρίπτεται. 160 καταπίπτει. Τροπολογία 9 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 που είναι ίδια με την 162, οπότε ψηφίζονται μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 163, υπέρ, κατά, αποχές, ξανά. Τροπολογία 163, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίθηκε. 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ε, βλέπω τι ψηφίζετε, τροπολογία 166, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 167. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 169. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της τροποποιημένης γνωμοδότησης με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Okay, Και τώρα περνούμε στον διαρθρωμένο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2018 Συστάσεις αναχώρα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τομπρόφσκης την Επίτροπο για την απασχόληση στα κοινωνικά θέματα, τις δεξιότητες, την κινητικότητα, κυρία Τίσεν, και τον κύριο Μοσκόβηση, ο οποίος όμως ζητεί συγγνώμη καθώς δεν θα μπορέσει να έρθει στον οικονομικό διάλογο σήμερα.